Αγαπητοί, συνάδελφοι, κυρίες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω με κάποια έκπληξη ότι είναι λίγες οι παρουσίες ε, στην αίθουσα και οι νυχτερινές συνεδριάσεις έχουν από ό,τι βλέπω κάποια παράλληλη αντανάκλαση σε αυτόν τον χρόνο ερωτήσεων που απευθύνονται προς το Συμβούλιο με την σπανίδα των παρουσιών. Αυτό είναι το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Ερωτήσεις λοιπόν προς το Συμβούλιο. Και περνάμε αμέσως ερωτήσεις μια και πιέζει πολύ ο χρόνος. Καλωσορίζουμε φυσικά τον κύριο Σαστέρ που εξ του Συμβουλίου παρίσταται ως Προεδρεύων θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση που θέτει ο συνάδελφός μας ε, κύριος Πόσελτ, Μπέρν Πόσελτ για την ταυτότητα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Έχει τον λόγο ο κύριος Πόσελτ λοιπόν. Παρακαλώ. Όχι, συγγνώμη. Για να απαντήσει ο κύριος Σαστέλ στην ερώτηση αυτή που υπέβαλε γραπτός ο κύριος Πόσελτ. Ο κύριος Σαστέλ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρο που μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του Συμβουλίου ενώπιον παρκούς ακροατηρίου στις θέσεις των επισκεπτών. Η ΕΠΑ, εκτός μικροφώνου σχόλια, θέλετε να θέσετε την ερώτησή σας όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρο. Η διαδικασία, κύριε Πόστολτ, είναι σαφή. Απαντά ο κύριο Αστέλ εξ ονόματο για την ερώτηση που θέσατε και κατόπιν θα έχετε την ευκαιρία να θέσετε περαιτέρω ερώτηση, συμπληρωματική κτλ. Το λόγο έχει ο κύριο Σαστέλ που θα απαντήσει στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως έλεγα, η ευρωπαϊκή πολιτική Άμυνα και ασφάλειας γνώρισε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη και έγινε ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία της ε, Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δέκα χρόνια περίπου μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής ε, ε, Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας που είναι κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και της κοινή πολιτική εξωτερικής πολιτική. η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ένας γνωστός παράγων στη διεθνή σκηνή. Οι πολλές αποστολές μας ανά τον κόσμο είναι απόδειξη. Κατόπιν πρωτοβουλία του Συμβουλίου και των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη ΕΠΑ έχει 24 αποστολέ σε τρει υπήρου πολιτικής, στρατιωτικής και στρατιωπολιτικής φύσεως. Η Ένωση είναι κατά συνέπεια παρούσα στο Αφγανιστάν, τη Γεωργία, την Μέση το Ιράκ, τη Σομαλία και στα, και στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι δεδομένο ότι η αποστολή αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση της ορατότητας της Ένωσης ε, στον τομέα αυτό. Το γενικό πλαίσιο των αποστολών αυτών περιγράφεται μεταξύ άλλων και από τη συνθήκη της Λισαβόνας που δίνει και το γενικό πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Σε ό,τι αφορά το Ευρωκόρπ, το, το Ευρωσώμα, υπενθυμίζω και το λέει και ο Πόσελ το ότι το, Ευρωσο, το Eurocorp δεν είναι τμήμα τη Ένωση, αλλά είναι ένα πολυ, πολυεθνικό χερσαίο στρατηγείο επιχειρησιακού χαρακτήρα. Γεννήθηκε το 1900 92 μετά από μια ιδέα του καγκελαρίου Κόλ και του Γάλλου Προέδρου ε, Μιτεράν έχει, ε, παρουσία, έχει παρουσία στο Κόσοβο και αλλού και έχει συμβάλει στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ε, ενόπλων δυνάμεων των των κρατών και την κοινή άμυνα και ασφάλεια. Ορισμένα κράτη της Ένωσης, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία μετέχουν στο, στο Eurocorp και πριν από λίγο καιρό το Europol άνοιξε και στην συμμετοχή άλλων κρατών μελών της Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η Προεδρία καταβάλει προσπάθειες στα πλαίσια της υλοποίησης της συνθήκης της Λισαβόνας και χαιρετίζουμε τη συμφωνία στα πλαίσια αυτά μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που θα αποτελέσει ένα μείζον εργαλείο για την αποτελεσματική υλοποίηση της, πολιτι... κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι η Βελγική Προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να επιτύχει μια συμφωνία με το Κοινοβούλιο στις τροποποιήσεις των δύο κανονισμών που συνδέονται στενά με την υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ό,τι αφορά το προσωπικό και το χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά τις, προεδρίες, τις, ε, τις πρωτοβουλίες της Προεδρίας στον τομέα της ΕΠΑ. Σας παραπέμπω στο πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας που αναφέρει ότι είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει στρατιωτικές και μη στρατιωτικές ικανότητες για να καλύψει τις αποστολές της, την διαθρωμένη και μόνιμη συνεργασία, την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Προγραμματισμού και διοίκηση των επιχειρήσεων κρίσεως, την ικανότητα ταχείας αντίδρασης και μια συνεκτική προσέγγιση, ιδίως στον τομέα ε, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας, κατάρτισης, διαχείρισης κρίσεων, ενίσχυση της Ευρωπαϊκής, Υπηρεσίας, ε, της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας και της στρατηγικής συνεργασίας Ένωσης και ΝΑΤΟ. Θέματα σημαντικά που απαιτούν ε, ιδιαίτερες προσπάθειες. Το Βέλγιο καταβάλει ιδιαίτερες ε, Πρωτοβουλίε σε ό,τι αφορά την ΕΠΑ και έχει οργανώσει πολλά σεμινάρια για θέματα δυναμικού, μόνιμης ε, διαθρωμένης συνεργασία και κατάρτισης. Όλα τα ζητήματα αυτά θα είναι στο κέντρο των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνα, αύριο και μεθαύριο στο Βέλγιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριε Υπουργέ. Κύριε έχετε μισό λεπτό για να διατυπώσετε την επερώτησή σας ή να συμπληρώσετε με ερώτηση, όπως θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα σύντομα μια παρατήρηση. Ήταν πολύ καλή απάντησή σας κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου προηγούμενα μόνο διαμαρτυρήθηκα για την κοινική παρατήρηση για τις παρουσίες. Όσοι έχουν διατυπώσει ερωτήσεις είναι παρόντες και δουλειά σας είναι να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους. Θέλω να πω σαφώς ότι η επερώτησή μου είναι η εξή. Σχεδιάζει το Βέλγιο μια πρωτοβουλία, αυτή είναι η ερώτησή μου, ώστε η κοινή εξωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια να προαχθεί. Έχουμε μια συζήτηση για την αναδιάρθρωση της, των ενόπλων δυνάμεων στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Θα ήταν μια ευκαιρία να αναλυφθεί πρωτοβουλία από πλευρά ε, του Βελγίου αντίστοιχα. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε κύριε Πόσετ. Θα λάβει τον λόγο ο κύριος Σαστέλ για να απαντήσει την επερώτησή σας. Κύριε Πόσετ. Πρόεδρε, να υπενθυμίσω προς τον κύριο Βουλευτή ότι στο τέλος της προηγούμενης παρέμβασής μου είπα ότι στο πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας υπήρχε μια σειρά ζητημάτων και θεμάτων που θα έπρεπε να ενισχύσουν την ε, συνεργασία μας, τη συνεργασία μας ιδιαίτερα στον τομέα, στον τομέα της άμυνας. Ότι το Βέλγιο έχει αφιερώσει πολλές πρωτοβουλίες σχετικά υπομορφή σεμιναρίων και συζητήσεων για θέματα δυνατοτήτων και σας παραπέμπω και στην επικαιρότητα. Την συζήτηση που θα ξεκινήσουν αύριο και μεθαύριο οι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Άμυνας που θα γίνει στην Γάνδη. Ευχαριστώ κύριε Σαστέλ. Ο κύριος Τσέμκε θέλει να υποβάλει μια συμπληρωματική ερώτηση όπως προβλέπει ο κανονισμός. Κύριε Ζέμκε έχετε το λόγο. Η, ερώτησή μου οφείλεται στο ότι ο Υπουργό είπε ότι αύριο και μετά αύριο θα γίνει άτυπη συνάντηση Συμβουλίου Υπουργών Άμυνα των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω να ρωτήσω το εξή. Εντό Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί μαχητικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά προς το παρόν. Ε, στις συζητήσεις θα τεθεί αυτό το ζήτημα ή θα, θα παραμείνουν θεωρητικές ή υπάρχουν και ομάδες κρούσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Κύριε Σαστέλ, θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση. παρόμοια με την προηγούμενη απάντηση έχω. Προφανώς θέλουμε να αυξήσουμε την δυνατότητα δράσης επιτόπου στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών αύριο, είναι προφανές ότι το ειδικό αυτό θέμα θα εξεταστεί. Θα δούμε τις επερχόμενες μέρες τι θα γίνει από την άτυπη συνάντηση των Υπουργών. Κάποιοι από αυτούς, όπως ξέρω, θέλουν να προχωρήσουν σχετικά. Ευχαριστώ. Να πω τα εξή στον κύριο Πόσελτ. Καταλαβαίνω ότι το ευγενικό σχόλιο του κυρίου Υπουργού, όπως το κατάλαβα τουλάχιστον εγώ, έρχεται σε συνέχεια του δικού σας, της δικής σας ε, παρουσίας ήταν ενδιαφέρουσα η ερώτηση, πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση και είναι κρίμα, και νομίζω όλοι πρέπει να το πούμε, που δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί συνάδελφοι στην αίθουσα. Γιατί στην ουσία χάνεται και η ερώτηση η δική σας και η απάντηση του κ. Υπουργού. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους. Δεύτερη ερώτηση της κυρίας Μακίνες και τρία του κυρίου Παπα-Νικολάου. Αποσύρθηκαν και οι δύο από τους συντάκτες. Η επόμενη ερώτηση που θα συζητήσουμε είναι η παριθμόν 4 της κυρίας Μπλινκεβιτσιούτε για τη μείωση της φτώχειας και του αποκλεισμού. Το λόγο έχει ο κύριος Σαστέλ για να απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας της κυρίας συναδέλφου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το, πρόεδρο... το πρόγραμμα του Συμβουλίου που συνέταξε το τρίο προβλέπει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και της ε, περιθωριοποίησης αποτελεί προτεραιότητα αφορά τα παιδιά, τις μονογονικές οικογένειες, τις ε, φτωχές οικογένειες. Και αυτά είναι κομμάτι της στρατηγικής ε, η Ευρώπης 2020 που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2010 από το Συμβούλιο που επίσης ενέκρινε την ε, συμπερίληψη του στόχου της, της φτώχειας και του αποκλεισμού αφαιρώντας από 20 εκατομμύρια άτομα ε, το φάσμα της φτώχειας μέχρι το 2020. Ένας άλλος στόχος είναι να ανεβεί στο 70% ε, η απασχόληση των γυναικών ε, της ενεργού ηλικίας και να μειώσει το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου. Στη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας θα ε, δώσουμε έμφαση σε τέσσερι θέματα. Το ελάχιστο ε, εισόδημα, κοινωνική προστασία, στέγη και κατάσταση των αστέγων, φτώχεια των παιδιών εντός των οικογενειών τους και τέλος συμμετοχή αυτών που είναι φτωχοί και όλων των εμπλεκομένων στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Προεδρία θα κάνει προσπάθεια να εμβαθύνει τη συζήτηση για το ελάχιστο εισόδημα στην Ευρώπη σε σχέση με τη φτώχεια. Η συζήτηση θα γίνει στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Στόχος είναι κάθε κράτος μέλος να εγκρίνει ένα ελάχιστο εισόδημα που θα εγγυάται ε, ένα επαρκές επίπεδο ζωής. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων η Προεδρία θα, αναγκαστεί, θα πιεστεί επίσης να προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη σημασία της αρχής της καλής διακυβέρνησης που συνεπάγεται ότι θα συμμετέχουν και αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση ένδυας. για να μπορέσουν όλοι να έχουν εγγυημένο δικαίωμα ε, στέγης, ασχολούμαστε με το θέμα της πρόσβασης της στέγης στη διάρκεια μιας ε, ε, διάσκεψη που θα γίνει 9 και 10 Δεκεμβρίου. Η Προεδρία θα θέσει σε προτεραιότητα το θέμα της φτώχειας των παιδιών και στην καταπολέμηση της κληροδότησής της από γενναία σε γενναία. Τέλος, η Βελγική Προεδρία στις 16 και 17 Δεκεμβρίου θα κλείσει το Ευρωπαϊκό Έτος της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού φροντίζοντας να ε, καταλήξει στα συμπεράσματα και στα διδάγματα για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Η συντάκτρια θέλει να κάνει μια επερώτηση. Έχετε μισό λεπτό να την θέσετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για μια απάντηση που κατανοώ πάρα πολύ καλά ότι είναι δουλειά των κρατών μελών να καταπολεμήσουν την φτώχεια και την, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Βελγική Προεδρία, κάθε επιτυχία ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αποφασίσουν τελικά όσον αφορά, αφορά το ένα ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα, κοινωνικό εισόδημα για τους πολίτες. Ποια είναι όμως η άποψή σας για την μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού. Επαρκεί για να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Σας ευχαριστώ κυρία. Ο κύριος Σαστέρ έχει τον λόγο να απαντήσει στην ερώτησή σας. Alors, si ma mémoire est bonne, Monsieur le Président, ε, αν δεν κάνω λάθος κύριε Πρόεδρε, εδώ και 15 μέρες εδώ στο, στην αίθουσα αυτή, στην ώρα των ερωτήσεων, απήντησα στην ίδια αυτή ερώτηση, επαναλαμβάνω ότι αυτή η μέθοδος είναι μια μέθοδος που πραγματικά μπορεί να ε, φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω αυτά που είπα, να, επα, να βεβαιώσω αυτά που είπα προ 15 μέρου. Σα ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Η ακόλουθη ερώτηση είναι εκείνη που διατυπώνει ο συνάδελφος μας κύριος Γκάλαχερ για το Διεθνές Συμπόσιο για την Επιστήμη και τις συμφωνίες για την αλληλεία. Έχει τον λόγο ο κύριος Σαστέλ, παρακαλώ. Euh, το συμπόσιο αυτό με τίτλο Διεθνές Συμπόσιο για την Βελτίωση Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Επιστήμης και Αλληλείας οργανώνεται από την Βελγική Προεδρία στις 9 και 10 Νοεμβρίου στην Οστάνδη. Πόλη, πολύ ωραία, παράκτια πόλη του Βελγίου όπως γνωρίζετε. Η Προεδρία έχει καλέσει άλλωστε και το Κοινοβούλιο όταν είχε παραστεί εδώ στις 15 για να παρουσιάσει τις προτεραιότητές του και θέλουμε με τα, στα πλαίσια του συμποσίου αυτού να συμβάλλει στις συζητήσεις για την προετοιμασία της μεταρρύθμισης της παρούσης κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Μια νέα κοινή πολιτική στον τομέα αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μετά το 2013 οι επιστήμονες και ο κλάδος της αλληλείας ε, συχνά έχουν διστάμενες απόψεις και ακολουθούν διαφορετικές θέσεις για την αλληλεία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ο στόχος του συμποσίου είναι να συζητήσει διεξοδικά το ζήτημα και να μάθει από τις βέλτιστες πρακτικές. Ε, προβλέπεται να οργανωθεί συζήτηση για πέντε θέματα, συλλογή δεδομένων και από αξιολόγηση αποθεμάτων, κοινέ προσπάθειε για τη βελτίωση τη επιλεξιμότητα και τη μείωση των απορρίψεων, επικοινωνία μεταξύ επιστήμων και κλάδου, βελτίωση των διαδικασιών ολοκληρωμένης ε, διαβούλευσης και εν τέλει η αυτοδιαχείριση. Τα αποτελέσματα του συμποσίου θα βοηθήσουν τη συζητή σε επίπεδο υπουργών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλίας του Νοεμβρίου κατόπιν το Συμβούλιο θα δράξει τα, συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργό. Έχετε 30 δευτερόλεπτα κύριε Γκάραγκερ για μια συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να συγχαρώ τον Υπουργό που κανόνισε αυτή τη σημαντική διάσκεψη και που συγκεντρώνει και τους επιστήμονες και τον τομέα της αλίας. Θέλω να τον ευχαριστήσω που δίνει έμφαση στο γεγονός ότι θα ε, δοθούν αποζημιώσεις για, για την... Για, την για τις απορρίψεις έτσι ώστε οι αλληλείς, γυναίκες και άνδρας θα ενθαρρυνθούν να φέρουν τη, το, τις ποσότητες αυτές στη στεριά. Και επίσης τα σκάφη κάτω από 15 μέτρα πρέπει να μπορούν να φέρουν εισόδημα επαρκές για να ζήσουν οι οικογένειές τους και να μην επηρεαστούν από τα νέα μέτρα. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Κύριε Σαστέρ, θέλετε να απαντήσετε στο σχόλιο αυτό στην κοινοβουλευτική παρέμβαση. Ευχαριστώ τον κύριο Βουλευτή για την πρότασή του. Τον ευχαριστώ και για τη... τους φόβους που εξέφρασε, τους μεταβιβάσεις, τον αρμόδιο υπουργό που θα προεδρεύσει του Συμποσίου. Επόμενη ερώτηση του κύριου Κρόλη για τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις Κροατίας στην Ένωση δεν θα συζητηθούν, θα συζητηθούν αλλά απόντος του κύριου Κράουλη θα την έχει αναλάβει ο κύριος Γκάραγκερ. Μπορείτε να απαντήσετε κύριε Σωστέλ. Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ένταξης με την Κροατία έχουν, έχουν προοδεύσει αρκετά, βρίσκονται στην τελική φάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρεται με τις σοβαρές προσπάθειες που έκανε η Κροατία στη διάρκεια του έτους αυτού και για την προόδο όσον αφορά την επίτευξη των κριτηρίων που έχουν τεθεί στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εν γέννη, στη φάση αυτή η διάσκεψη ένταξης ε, ε πρόκειται να ανοίξει 30 και 30, κεφάλαια 30 και 35 και να κλείσει 23. Ε, λόγω της μεγάλης προόδου η Κροατία πρέπει να συνεχίσει αυτή την δυναμική μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως είναι η δημόσια διοίκηση η ε, δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία των μειονοτήτων, η επιστροφή των προσφύγων, η δίωξη των ε, ε, που έχουν σχέση με τα εγκλήματα πολέμου και ε, πολλούς άλλους τομείς. Η Βελγική Προεδρία, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της, είναι αποφασισμένη να βοηθήσει την Κροατία να πραγματοποιήσει καθοριστική πρόοδο διαπραγματεύσεις, κλείνοντας το ταχύτερο δυνατόν τα περισσότερα και δυνατά κεφάλαια και υπό την έννοια αυτή είναι απαραίτητο η Κροατία να ολοκληρώσει τις ε, μερθαριθμίσεις του τομεί που ανέφερα και να ικανοποιήσει το, των, το σύνολο των κριτηρίων που παραμένουν εντός των προθεσμιών και συγκεκριμένα τα κεφάλαια που πρέπει να εξετάσουν τα κράτη-μέλη και που ενδεχομένως μπορούν να ολοκληρωθούν, να κλείσουν εάν θεωρηθεί ότι οι παράμετροι κλεισίματο έχουν τηρηθεί από την Κροατία είναι τα εξή πολιτική ανταγωνισμού και, ε, ε, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, αλληλεία, ε, περιφερειακή πολιτική και συντονισμό των διαρθρωτικών μέσων δικαστικές αρχές και θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιοσύνη, ελευθερία, ασφάλεια, περιβάλλον, εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας και δημοσιονομικές και ε, ε, χρηματοοικονομικές διατάξεις. Τρία κεφάλαια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο, επιτάπητο στο Συμβούλιο για ε, προσωρινή προσωρινό κλείσιμο, ελευθερία κεφαλαίων και κρίση κεφαλαίων, πολιτική μεταφορό και τέλος τα διάφορα, το 30, κεφάλαιο 35 πρόκειται να, να εξεταστεί ε, σε ένα μετέπειτα στάδιο. Κύριε Κάραχερ, θέλετε να υποβάλλετε συμπληρωματική ερώτηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Υπουργό για τα, την πληρέστατη απάντησή του. Να ρωτήσω το εξής μπορεί να με ενημερώσει αν, ή να μου το πει αν δεν το ξέρει τώρα. Πότε θα όταν... ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και χρειαστεί να ληφθεί η απόφαση, η απόφαση θα ληφθεί μόνο από το Κροατικό Κοινοβούλιο ή θα μπορέσει και ο λαός της Κροατίας μέσω δημοψηφίσματος να αποφασίσει για το μέλλον της χώρας. Ευχαριστώ κύριε Γκάλαχερ. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή. Πρόφανως είναι δικό μας θέμα να κρίνουμε την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί επιτόπου στην Κροατία. Μπορώ να καθορίσω ένα χρονοδι... Ε, διάγραμμα μόνο ανάλογα με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Κροατία, αλλά στο τέλος αυτής της διαδικασίας, μετά από επαφές ε, και ανταλλαγές με τον Κροάτη συναδερφό μου, προβλέπεται ότι τελικά ο λαός Κροατίας θα ε, γνωμοδοτήσει, θα, εκφράσει τη γνώμη του για την ένταξη. Ε, Κύριε Ζέμκε, θέλετε εσείς να θέσετε μια συμπληρωματική ερώτηση. Έχετε το δικαίωμα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια ερώτηση που θεωρώ σημαντική. Είπατε κύριε Υπουργέ ότι από τα 35 κεφάλαια έχουν ξεκινήσει τα 33. Περιγράψατε την πρόοδο στα 33. Εγώ έχω διαφορετική ερώτηση. Ποια είναι αυτά τα δύο που δεν έχουν ανοίξει. Αυτό είναι βασικό για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξέρετε κύριε Σαστέλ. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω ιδέα. Θα σας απαντήσω γραπτός. Θα απαντήσω στο αξιότιμο βουλευτή αμέσως. Έχω, δεν ξέρω απ' έξω τα 35 κεφάλαια, ποια μόλις ανοίξαν, ποια κλείσαν, ποια πρόκειται να κλείσουν, ποια δεν θα ανοίξουν. Νομίζω ότι απήντησα εξαντλητικά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κάθε κεφάλαιο. Αν δύο από αυτά δεν έχουν ανοίξει, ε, θα σας τα στείλω γραπτός. Σίγουρα κύριε Σαστέλ ε, θα είναι ικανοποιημένο ο κύριος και αν του στείλετε γραπτή απάντηση. Σύντομα. Ερώτηση 7 της κυρίας Χάρκιν. Δημογραφία και φροντιστές. Άτομο που παρέχουν φροντίδα στο σπίτι δηλαδή. Κύριε Υπουργέ. Monsieur le euh, euh, Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Βουλευτή έδωσε, έθεσε μια πολύ ανησυχητική ερώτηση αυτή την δύσκολη οικονομική περίοδο. Καταλαβαίνουμε το κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα άτομα που κάνουν θελοντική δουλειά και που υποχρεούνται τώρα να μην κάνουν τόσο πολύ για να ψάχνουν δουλειά. Το ζήτημα αφορά την επανένταξη των ατόμων αυτών στην αγορά εργασία. Το Συμβούλιο έχει επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίσουν τα άτομα αυτά που διέκοψαν την καριέρα του για να αναλάβουν ευθύνε μη αμοιβόμενη βοήθεια και ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν ούτω ώστε οι περιπτώσει των ατόμων αυτών να λαμβάνονται υπόψη στη στα συνταξιοδοτικά καθεστώτα, στην οδηγία για την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαίσιων για την γονική άδεια, το Συμβούλιο τόνισε ότι μετά την έκβαση της γονικής άδειας ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επανέλθει στη θέση εργασίας του ή να βρει μια ισοδύναμη ή αντίστοιχη εργασία ε, βάσει του παλαιού συμβολέου. Το Συμβούλιο ξέρει ότι οι κοινωνικοί εταίροι που έδωσαν την άποψη ε, του στην Επιτροπή για το νέο τύπο οικογενειακής άδειας όπως άδεια για φροντίδα μέλους οικογένειας πρέπει να, λαμβάνουν υπόψη και τη δεύτερη διάσταση καλύπτει και τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η ανάληψη τη ευθύνη τη οικογένεια ανήκει εμπολή ακόμα στην ε, γυναίκα λόγω των ε, κοινωνικών στερεοτύπων, κυρίω ό,τι αφορά τον ρόλο άνδρα και γυναίκα στην κοινωνία. Στο πλαίσιο του προγράμματος δράση του Πεκίνου, το Συμβούλιο υιοθέτησε ήδη από το 2007 συμπεράσματα για το ζήτημα των γυναικών και τη φτώχεια με μια σειρά δικτών που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη και την Επιτροπή να παρακολουθήσουν το βασικό αυτό ζήτημα. Στα συμπεράσματα του το Συμβούλιο χρειάστηκε να καταλάβει και έδειξε ότι έχει επίγνωση πως η ανάληψη μη αμοιβόμενη δραστηριότητα αντί για αμοιβόμενη μπορεί να αποτελέσει προσωπική επιλογή. Αλλά ότι λόγω των ανισοτήτων μεταξύ φύλων ε, είναι ένα πρόβλημα πολύ ειδικό για τις γυναίκες που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική τους εξαρτησία και το επίπεδο κοινωνικής τους προστασίας ιδίως στη φάση της συντάξεως όταν πολλές γυναίκες μπορεί να χρειαστεί, χρειάζεται μάλλον να μείνουν με πολύ μικρές συντάξεις. Υπό την οπτική αυτή το Συμβούλιο δήλωσε ότι χρειαζόταν να υπάρξει πιο δίκαιη κατανομή των βασικών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών και τόνισε την ανάγκη βελτίωσης των υποδογμών υποδοχής παιδιών, τη δημιουργία ε, θεσμών ενίσχυσης άλλων κατηγοριών πληθυσμού και ότι κάτι τέτοιο σημαίνει πως ο αριθμό των ανθρώπων, ενώ η γύρανση του πληθυσμού σημαίνει ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που θα χρειάζονται βοήθεια και ότι η, η ισότητα μπορεί να βοηθήσει την ε, απασχόληση. Και γι' αυτό το 2009 υπογράμμισε τη σημασία μακροπρόθεσμα της προσέγγισης αυτής για την Ένωση, συμπεριλαμβάνοντας και την δημογραφική διάσταση, καθώς και τον συσχετισμό μεταξύ υψηλής απασχόλησης των γυναικών και υψηλών ποσοστών γονιμότητας. Γι' αυτό το Συμβούλιο πρότεινε την υιοθέτηση πολιτικών που θα επιτρέπουν και, στο γυνα... και στη γυναίκα και στον άνδρα την καλύτερη... το συγκαλύτερο συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματική ζωής. Κυρία Χάρκιν, θέλετε να συμπληρώσετε το ερώ... την ερώτησή σας. Ε, ε, ναι, βεβαίω. Ευχαριστώ για την πολύ ολοκληρωμένη απάντηση, κύριε Υπουργέ. Είναι προφανέ ότι το Συμβούλιο αντιμετωπίζει το θέμα με σοβαρότητα και με ενδιαφέρει να ακούσω ότι ε, μελετάτε το θέμα της οικογενειακής άδεια. Είναι είναι τα στάνταρ που ισχύουν για αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν. Επίσης αναφερθήκατε και στο σκέλος του φύλου. Επίσης, πολλοί νέοι άνθρωποι καταλήγουν να φροντίζουν ηλικιωμένους και αυτό το ξεχνάμε και αναφερθήκατε στην προσωπική επιλογή. Αυτό θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ε, θέλουν να έχουν την επιλογή να μπορούν να προσφέρουν αυτή τη φροντίδα ή όχι. Και επίσης χαίρομαι που λάβατε υπόψη σας και το θέμα των συντάξεων γιατί οι άνθρωποι αυτοί χάνουν ένα μέρος του μισθού τους, δεν μπορούν να κάνουν χάνουν κοινωνικές εισφορές λόγω αυτής της φροντίδας που προσφέρουν και χάνουν συντάξεις. Ίσως λοιπόν είναι κάτι, ε, ένας τομέας όπου θα μπορούσε το Συμβούλιο να κάνει συστάσεις στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Υπουργός μήπως θέλει να απαντήσει στην, περαιτέρω ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά η κυρία επανέφελαβε αυτά που είπα στην απάντησή μου και πραγματικά συμφωνώ μαζί της κυρίως για αυτές που κάνουν επιλογή ζωής δεν πρέπει να τιμωρηθούν στο τέλος της καριέρας τους, θα πρέπει να μπορούν να χαρούν μια αξιοπρεπή σύνταξη και αυτό είναι ο σκοπός του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή. Η επόμενη ερώτηση στη σειρά που έχουμε είναι της ε, κυρίας ε, Τσίσκα που υιοθετήθηκε από τον κύριο Βαλένσα τι απουσία του συναδέρφου αναφέρεται σε σχέση με τις εκπομπές ε, του σταθμού Αλάξα. Έχετε τον λόγο για να απαντήσετε κύριε Σαστέλ παρακαλώ. Τη 10 Μαρτίου του 2010 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν την οδηγία 2013 για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης που καθορίζουν το πλαίσιο παροχής οπτικοακουστικών μέσων στην Ένωση. Το άρθρο 6 προβλέπει τα κράτη-μέλη φροντίζουν με κατάλληλα μέτρα επειδή οι υπηρεσίες των οπτικοακουστικών μέσων που παρέχουν ε, την αρμοδιότητά τους να μην παρέχουν καμία υποκίνηση προς μίσος με βάση το, τη θρησκεία, το φύλλο ή ε, την εθνικότητα. Επίσης πρέπει να φροντίσουν τα κράτη-μέλη να φροντίσουν την εφαρμογή της οδηγίας και η Κομισιόν ως ε, θεματοφύλακα των συνθήκων να φροντίσει για αυτό επίσης. Επίσης, σύμφωνα με, το, ε, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει τα κράτη να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητά τους αν χρησιμοποιείται δορυφόρος που έχει σχέση με το κράτος μέλος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρει το αξιότιμο μέλος, το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται ότι η Κομισιόν έθεσε το θέμα στη, σε γνώση των αρμόδιων γαλλικών αρχών, της ΕΣΑ, οι οποίες αυτή τη στιγμή το εξετάζουν. Δεν είναι λοιπόν θέμα του Συμβουλίου να σχολιάσει την έρευνα αυτή η οποία είναι εν εξελίξη. Σα ευχαριστούμε κύριε Βαλένσα. Θέλετε να κάνετε μια συμπληρωματική ερώτηση, μια περώτηση, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα συμφωνούσα, πρέπει να πω, με το τελευταίο τμήμα τη απάντηση του κυρίου Σαστέ. διότι θεωρώ ότι είναι στι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου να προσέχουν ιδιαίτερα τέτοιε επανειλημμένε και αρνητικέ τάσει στην λειτουργία αυτού του τηλεοπτικού σταθμού και δορυφορικά είναι μια άλλη στιγμή και πρέπει να ξέρει κανείς ε, ότι ξαναστέλνουν αυτές ε, μέσω των ε, εκπομπών τους αυτά τα μηνύματα. Παρακάμπτουν την νομοθεσία. Και αυτό το θέμα ακριβώς η ερώτησή μας εκφράζει την ανησυχία μας. Τι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτό το κρυφτούλι να σταματήσει επιτέλους. Σας ευχαριστούμε κύριε Βαλένσα. Θέλετε να σχολιάσετε κύριε Σαστέλ παρακαλώ. εν μέρη συμφωνώ με την ερμηνεία σας. Βεβαίως τα κράτη-μέλη ελέγχουν την Κομισιόν για την τροποποιήσει της οδηγίας στο Συμβούλιο και οι συνομοθέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εν μέρει μια ευθύνη γιατί έχουν θέσει, ε, έχουν δημιουργήσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, αυτό που αναφέραμε, και τα κράτη-μέλη που τον έλεγχο της Κομισιόν πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή αυτή την οδηγία. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαστέρ. Τώρα συνεχίσουμε σε σχέση με τις ερωτήσεις και βλέπω ότι και για την ερώτηση 9 και για την 10 από πλευράς της κυρίας Τίκαου και που ο κύριος Ταραβέδα είχε, την είχε αναλάβει την απουσία και η ερώτηση 10 του συναδέλφου Σον Κέλλη αποσύρθηκαν τη απουσία εκείνων που θα τις διατύπωναν. Στη συνέχεια έχουμε την ερώτηση 11 που, θα που διατυπώνει ο κύριος Όλε Σμιτ για την κατάσταση της μειοψηφίας των Ρωμάτων συγκάνων στην Ευρώπη και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σαστέλ, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση του κύριου Σμιτ. Κύριε Πρόεδρε, μετά τη δεύτερη διάσκεψη κορφής της Ευρώπης για τους Ρωμά που έγινε στο Κορτού τον Απρίλιο, στις 18 ε, Ιουνίου 2010 τα συμπεράσματα λέει πρέπει να προχωρήσει η κατάσταση των Ρωμά ε, και ένα μεγάλο ποσοστό των Ρωμά βρίσκεται σε καταστάσεις εξαιρετικής ένδυας, υφίσταται διακρίσεις και αποκλεισμό, πράγμα που σημαίνει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ανεπαρκή συνθήκες διαβίωσης, ανεπαρκή ε, πρόσβαση στην εργασία και υγειονομικές συνθήκες. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρώμα με βάση την απόφαση αυτή και τις συστάσεις που διατύπωσαν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εγγυόμενοι την καλύτερη δυνατή και αποτελεσματικότερη προσφυγή στα υφιστάμενα μέσα. Το Συμβούλιο επίσης υπογράμμισε τη σημασία να φροντίσουμε την ενεργο... για την ενεργό συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών ε, αρχών και των ίδιων ρωμάτων, το Συμβούλιο της Στοχόλμης και το, το, το πρόγραμμα της Στοχόλμης και το Συμβούλιο ε, ε, αναφέρει ε, στα συμπεράσματά του συγκεκριμένα τους Ρώμα και ζητά την, της, να γίνει προσπάθεια για να ενταχθούν στην κοινωνία οι ευάλωτες ομάδες. Τα μέτρα που πρόσφατα ένα κράτος μέλος έλαβε σε σχέση με άτομα που ανήκουν στους Ρώμα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στη διάρκεια του γεύματος του, Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16 Σεπτεμβρίου και ο πρόεδρος ανακοίνωσε τη συνένεση που προέκυψε από αυτή τη συζήτηση με τα τρία σημεία. Ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα να πάρει μέτρα για να γίνει σεβαστό το δίκαιο στο εδαφός του. Η Κομισιόν έχει το δικαίωμα ή μάλλον το καθήκον να φροντίζει να τηρεί το δίκαιο από τα κράτη-μέλη και στην επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα Τη της ενσωμάτωσης των Ρώμα θα συζητηθεί. Επιπλέον, η Προεδρία η Βελγική Προεδρία ε, διατύπωσε την ευχή η κατάσταση των Ρώμα να τεθεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου έπσκος 21 Οκτωβρίου. Το Συμβούλιο αυτό δεν θα συζητήσει τα αποτελέσματα της άτυπης συνάντησης που έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι και που κατά την άποψή μου, εξ όσων γνωρίζω, δεν αφορούσαν συγκεκριμένα την κατάσταση των Ρώμα. Σας ευχαριστούμε. Κύριε, κύριε Σμιτ, θέλετε να κάνετε μια επερώτηση. Έχετε δικαίωμα να παρέμβετε για μισό λεπτό, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για την απάντησή σας. Θα ήθελα να πω Ευχαριστώ. Έχετε εσείς την δυνατότητα και από των 27 κρατών μελών άμεσα να αντιδράσετε. Είναι μια δυσχερή κατάσταση για την Ευρώπη. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά Τσιγκάνοι επί αιώνε διώκοντο. Κατά το τελευταίο διάστημα καταδείχθηκε σαφώ ποιε ελλείψει υπάρχουν στην Ευρώπη. Πώ θέλουμε να επεξηγήσουμε σε άλλε χώρε πώ πρέπει να φέρονται όταν εμεί δεν φερόμαστε σωστά, ενώ θα έπρεπε. Και από πλευρά δημοσιογράφου και συγγραφέω που έχει γράψει ένα βιβλίο «Θάψτε με όρθιο» Και ε, σε σχέση με αυτό το θέμα, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να παρακαλέσω το Συμβούλιο από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει μια επιτροπή για τη διαπίστωση τη αλήθεια, τη διακρύβωση τη αλήθεια. Να δει τι έγινε στην ευρωπαϊκή ιστορία με του Ρωμά, με του Τσιγκάνου. Είναι αναγκαίο να εξετάσουμε το ιστορικό παρελθόν, γιατί δεν μπορούμε κατά άλλα να είμαστε αξιόπιστοι αν δεν το κάνουμε. Σα ευχαριστώ θα έχετε το δικαίωμα για ε, το μισό λεπτό που χρησιμοποίησατε ήταν το μεγαλύτερο όλη τη ε, χρονομέτρηση. Έχετε τον λόγο, κύριε Σαστέρ, για να απαντήσετε. Καταγράφω την πρότασή σα να επαναξετάσουμε την ιστορία μας για το ζήτημα αυτό. Και να σας πω επίσης ότι σε ένα ζήτημα που είναι γεγονό ότι ήταν ιδιαίτερα θερμό τις τελευταίες εβδομάδες, ότι το Συμβούλιο που εκπροσωπώ σήμερα περιμένει πολλά από την Επιτροπή, ιδίω την λεπτή ανάλυση του θέματο, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση τη επικαιρότητα που βιώσαμε τι τελευταίε εβδομάδε. Δεν είναι λοιπόν αρμοδιότητα του Συμβουλίου να κρίνει την α ή β κατάσταση, αλλά της Επιτροπής να μα πει κατά πόσον η συνθήκη και οι οδηγίε τηρήθηκαν επί του στήματος αυτού. Σας ευχαριστούμε. Η ερώτηση 12 της κυρίας Ρόδη Κράτσα για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και της ψηφιακής αγοράς καταπίπτει τη απουσία της συντάκτριας και περνάμε στο 13. Ερώτηση 13 του συναδέφου Jim Higgins για το εμπόριο παιδιών. Παρακαλώ. Σαστέλ, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Η υφιστάμενη νομοθεσία για την πρόληψη και καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων περιλαμβάνει κατά βάση μια απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου τη 19η Ιουλίου του 2002 για την καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη ιδίω να επιβάλλουν κυρώσεις και να καταστήσουν ποινικά δικήματα την εκμετάλλευση ανθρώπων για την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική ή επαγγελματική εκμετάλλευση. Οι πρώτες οδηγίες για την καταπολέμηση της, της ε, εμπορία παιδιών και την προστασία των, των θυμάτων και μια δεύτερη οδηγία για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και τη παιδική πορνογραφία βρίσκονται υπό εξέταση αυτή τη στιγμή στα πλαίσια των, εργών, των οργάνων της Ένωση. Οι προτάσει αυτές έχουν στόχο την υιοθέτηση ειδικών μέτρων προστασίας ε, και βοήθειας σε παιδιά που είναι θύματα εμπορία ανθρώπων. Περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις για την βελτίωση των διώξεων πράξεων που διαπράττονται εκτός επικράτειας της Ένωσης και κανόνες εν της πρόληψη, για την πρόληψη τέτοιων ε, ε, αδικημάτων. Με βάση το πρόγραμμα της Στοκόλμης δίδεται ειδική ε, προσοχή στα παιδιά που είναι ιδιαίτερα τροτά, ιδίως παιδιά θύματα εκμετάλλευσης και σεξουαλική σεξουαλικών καταχρήσεων και παιδιά που είναι θύματα εμπορία ασυνόδευτοι ανήλικοι στα πλαίσια της πολιτικής μετανάστευση τη Ένωση. Πρέπει επίση να προσθέσουμε ότι η Επιτροπή υιοθέτησε ένα πρόγραμμα δράση για του ασυνόδευτους ανηλίκους που προτείνει μια κοινή προσέγγιση που θα βασίζεται στην αρχή του απότερου συμφέροντος του παιδιού και την, ε, μια σειρά δράσεων όπως η πρόληψη, η υποδοχή, η βιώσιμη προστασία και μετά από τις προτάσεις αυτές το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του για τα ασυνόδευτα ανήλικα που υιοθέτησε τον Ιούνιο του 2010 ζήτησε από τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων αναθέτοντας τα παιδιά αυτά στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Είναι δύσκολο τώρα να ορίσουμε πόσα ακριβώς είναι, πόσα άτομα είναι θύματα εμπόδια ανθρώπων εκτός της Ένωσης. Η ατόμων που μπαίνουν παράνομα στην Ένωση στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων και με στόχο να παράσχουμε στην Ένωση αντικειμενικές και αξιόπιστες συγκρίσιμες στατιστικές το Συμβούλιο θέτησε στα συμπεράσματα του Ιουνίου του 2009 για την ε, θέσπιση, την θέσπιση ενός άτυπου ε, πλαισίου εθνικών εισηγητών ε, για ε, ενός δικτύου, άτυπου δικτύου ε, ειδικών εισηγητών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενώ δημιουργήθηκε και μια δομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, ένα κείμενο γενικής, γενικού προσανατολισμού για την αντιμετώπιση τη εμπορία παιδιών υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2009 και τμήμα του περιλαμβάνει το ζήτημα τη εμπορία παιδιών. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που αφορά συγκεκριμένο κράτο μέλος ε, δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου να λαμβάνει θέση επί συγκεκριμένων ερωτημάτων. Κύριε Χίγκιν, θέλετε να κάνετε μια συμπληρωματική ερώτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η διακίνηση των ανθρωπίνων όντων είναι το χειρότερο έγκλημα, αλλά η παράνομη διακίνηση ενηλίκων είναι κάτι το φοβερό. Αλλά για τα παιδιά είναι ακόμα χειρότερο. Όσον αφορά τη χώρα μου, ξέρω ότι έχουμε την νομοθεσία του 2002. Έχουμε ε, αρκετά άσχημα αποτελέσματα 441 ε, ε, παιδιά ε, λείπουν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αποτελεσματική δουλειά η οποία θα μπορέσει να σταματήσει μια για πάντα αυτή την παράνομη διακίνηση γιατί υπάρχουν ανοιχτά σύνορα πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε σοβαρά και πραγματικά χαίρομαι που το Συμβούλιο έχει τέτοια αποφασιστικότητα. Σα ευχαριστούμε κύριε Higgins. Κύριε Σαστέρ θέλετε να αντιδράσετε στο σχόλιο του κυρίου Higgins παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω το αξιότιμο μέλος για τα όσα είπε σε σχέση με το Συμβούλιο και να επαναλάβω ότι πράγματι η βοήθεια και η προστασία των ε, θυμάτων είναι βασική ε, βασικό στόχος της οδηγίας για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και το Συμβουλίο θα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει αυτό το θέμα ε, τη δημιουργία του αποτελεσματικού δικτύου και να μπορέσει να πείσει τα κράτη-μέλη να αναλύσουν τις βέλτιστες πρακτικές όπου και αν εφαρμόζονται για να εναρμονιστούν όλοι οι σχετικοί κανόνες. Σας ευχαριστούμε. Η ερώτηση 14 και που είχε καταθέσει ο συνάδελφος Λέαμ Έργοντ για την Ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά μέτρα για την δημιουργία θέσεων εργασίας την έχει αναλάβει ο κύριος Γκάλαγκα και έχει σπάσει το ρεκόρ όπως καταδεικνύεται στην ε, παρουσίαση ερωτήσεων εξ των συντακτών. Έχει τον λόγο ο κύριος Σαστέρ τώρα για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Παρακαλώ. Κύριε Γκάλαχερ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Τα κράτη-μέλη είναι κυρίω αρμόδια όσον αφορά τον καθορισμό και την υλοποίηση τη εθνική πολιτική σε θέματα απασχόληση, δεδομένου ότι η κατάσταση τη αγορά εργασία διαφέρει από κράτο σε κράτο. Τα μέρα που πρέπει να ληφθούν, κατά ανάγκη, διαφέρουν όμως, συνολικά συνεισφέρουν στην επίτευξη των συνολικών στόχων της Ένωσης. Με βάση τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα συντονίζονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης που προβλέπει μεταξύ άλλων κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Ιουνίου 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Γενική Κατεύθυνση των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών για την ενσωμάτωση των, της οικονομικής πολιτικής και της απασχόλησης που αποτελούν βασικό στοιχείο της υλοποίησης στρατηγικής 2020 για την απασχόληση και την ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου της 8 η Σεπτεμβρίου 2010, η Προεδρία θα υποβάλει ε, τα συμπεράσματα αυτά στο Συμβούλιο προσέγγιση την, την επόμενη συνεδρίαση του ΕΠΣΚΟ στις 21 ε, Οκτωβρίου 2010. Οι κατευθυντές αυτές γραμμές προβλέπουν ότι τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσουν μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια μιας ευφυού βιώσιμης και ε, ε, ανάπτυξης που να συμπεριλαμβάνει τους πάντες με σκοπό τη βελτίωση κατάστασης στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα για τις ομάδες που υποεκπροσωπούνται οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, αυτοί που έχουν λίγα ε, προσόντα, οι νόμιμοι μετανάστες να ε, βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά της διαρθρωτικής ανεργίας και να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην ζήτηση και την προσφορά. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εργατικό δυναμικό που να έχει τα προσόντα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει, να μπορέσει να προωθηθεί η διαβίου ε, μάθηση και να δημιουργούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα κατάλληλο Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους και να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόσβαση στην απασχόληση και στην αγορά αγορά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα στις μειονεκτικές περιοχές και μέσα των κοινών εκθέσεων ε, για την απασχόληση. Το Συμβούλιο μαζί με την Κομισιόν παρακολουθεί κατάσταση απασχόληση στα κράτη-μέλη και κυρίως την υλοποίηση των καθηγητήρων γραμμών για την απασχόληση ε, και την κοινή έκθεση για την απασχόληση 2009-2010, το οποίο πιστά ε, απεικονίζει τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η κατάσταση στην απασχόληση και κυρίως την απασχόληση των νέων και των γυναικών. Παραδείγματο χάρη το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιώσουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων, να υποκινήσουν τη θέση, δημιουργία θέσεων εργασία πράσινη και να βοηθήσουν τι επιχειρήσει να εξυγχρονίσουν τη βιομηχανική του βάση δεδομένη τη σημαντική τη σημασία τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Συντονισμού τη Απασχόληση ε, και να για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής η οποία έχει σημαντικό ε, ρόλο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Σε ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κύριε Γκάλαγερ, η επερώτησή σας παρακαλώ. Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την απάντηση. Παρότι τα σχέδια είναι πολύ Ωραία. Πιστεύω ότι να μπορούν να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχτηκε ότι η Ευρώπη έχει έλλειμμα στη μια 1,5 εκατομμύρια θέσεων εργασία άμεσα και υπάρχει υπερβολική νομοθεσία απασχόλησης. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στις εθνικές πολιτικές όμως θα θυμόσαστε ότι στην ομιλία του κ. Μπαρόζο για την κατάσταση της Ένωσης αναφέρθηκε στην ε, απόφασή του να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία. Ποια είναι η άμεση δράση που μπορεί να αναλάβει το Συμβούλιο να εξασφαλιστεί ότι αυτή η γραφειοκρατία θα περιοριστεί και θα αυξηθούν θέσεις εργασίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκάλαχερ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ για να απαντήσετε. Σα παραπέμπω ευθύ εξ αρχή το πρόγραμμα τη Βελγική Προεδρία επ' αυτού, γιατί το θέμα τη απασχόληση. Ε, περιλαμβάνεται στα διαρθρωτικά μέσα που αφορούν την απασχόληση μέσω της στρατηγικής του 2020. Βεβαίως όμως έχετε απόλυτο δίκιο στο βελγικό πρόγραμμα έχουμε μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στη μείωση του διοικητικού άχθους πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικροεπιχειρήσεις που δεν έχουν την διαρθρωτική ικανότητα να αποκτήσουν προσωπικό για να αναλύουν το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα όλα όσα αφορά τις ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις που είναι πάρα πολύ σύνθετα για τις μικρές επιχειρήσεις. Γι' αυτό γνωρίζω ότι στο Βέλγιο και τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας ο αρμόδιος υπουργός ε, σκοπεύει με βάση μια άτυπη διάσκεψη που οργανώνει να δώσει έμφαση σε, αυτή την, σε αυτό το ε, διοικητικό άχθο, σε αυτό το πρόβλημα που εμποδίζει την καλή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Μας πληροφορούν ότι ο κύριος Άλαν έχει αποσύρει την ερώτηση του υπαριθμού 15. Εκείνη της κυρίας Αντρικένε, η 16, καταπίπτει την απουσία της συντάκτριας και η 17 του κυρίου Ρίτσαρντ Χόουιτ για τις προόδους σε σχέση με την οριζόντια οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων υιοθετείται ότι η απουσία της, του συντάκτη από την κυρία Κίνγκα Έχει τον λόγο ο κύριο Σαστέρ για να απαντήσει αυτή την ερώτηση μετά από την παρέμβαση της κυρίας Γκέντς le memorandum d'entente auquel το μνημόνιο συνεννόησης ε, στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Βουλευτής. Είναι η ερώτηση 17, κύριε Υπουργέ. Alors, au cours de la présidence espagnole. Κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας, το Συμβούλιο συνέχισε την εξέταση της πρώτη οδηγίας και στις 7 Ιουνίου του 2010 σημείωσε μια έκθεση της Προεδρίας για την πρόοδο των εργασιών. Σύμφωνα με την έκθεση, θα είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η διεξοδική εξέταση της πρότασης, ιδίως ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις διατάξεις για την αναπηρία, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Τα μέλη του Συμβουλίου επέμειναν επίσης ως προς την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου όσο μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου γίνεται και ταυτόχρονα η αρχή της επικουρικότητας. Η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της συνθήκης ε, λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που απαιτεί ομοφωνία των μελών του Συμβουλίου. Αν το σχέδιο οδηγία ε, ε, έχει στόχο την επίτευξη ορισμένων από του στόχου τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίε, το εργαλείο αυτό δεν έχει ωστόσο στόχο να υλοποιήσει νομικά τη Σύμβαση, που έχει μια εκτενέστερη αρμοδιότητα από αυτέ των αρμοδιοτήτων τη Ένωση. Είναι αυτονόητο τόσο ότι ένα από του στόχου των συζητήσεων που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο έχουν να κάνουν με την συνέπεια και την συνοχή με τη σύμβαση αυτή. Αλλά και σε ό,τι αφορά το, το οικονομικό κόστος της ισότητα, οι συζητήσει αφορούν το, την έννοια του δυσβάστακτου βάρου του δυσανάλογου βάρους και την προσπάθεια να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ ε, πρόσβασης και οικονομικού κόστους της πρόσβασης. κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε ομοφωνία, βεβαίως το Συμβούλιο ωστόσο δεν είναι σε θέση να προβλέψει την έκβαση και τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Η κυρία Γκέντς παρακαλώ για μια ερώτηση. Έχετε τον λόγο τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας αναφέρω, Πρόεδρε, ότι προσπάθησα να κατανοήσω καλύτερα ποια επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα υπήρχαν από πλευράς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση και με το 2008 και γι' αυτό υπάρχει αυτό το θέμα που έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του χρόνου το Ευρωπαϊκό, ε, το, έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την, το επόμενο έτος μια ε, οδηγία. Υπάρχει ευθύνη φυσικά σε σχέση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν κύριε Σαστέ, βλέπετε εδώ κάποια δυνατότητα ώστε στο άμεσο μέλλον, προσεχώς, μετά την ανάλυση των προϋποθέσεων αυτών, να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το θέμα. Νομίζω η κρίση αυτή ήταν μια προειδοποίηση. Μια προειδοποίηση ότι τα ίσα δικαιώματα είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι η κρίση έχει καταστήσει την δυσχερή κατάσταση ακόμα δυσχερέστερη για τους πολίτες. Έχει τον λόγο κύριο Αστέρ για να απαντήσει παρακαλώ. καταλαβαίνω αυτά που είπε η κυρία Βουλευτής και τις προθέσεις ε, ε, για το ζήτημα. Προφανώς όντω είναι γεγονός ότι μπορεί να καθυστερούν οι συζητήσεις, αλλά πρόκειται για καινοτόμο κείμενο με τεράστιες ε, επιπτώσεις πρακτικού χαρακτήρα και παραλαμβάνω ότι απαιτείται ομοφωνία από τα κράτη-μέλη και συνένεση του Κοινοβουλίου για να εγκριθεί η οδηγία. Οι διεξάγονται αυτή τη στιγμή σύνθετες περίπλοκες συζητήσεις στο Συμβούλιο στην ομάδα εργασία ε, για κοινωνικά θέματα που έχει ήδη συζητήσει την πρόταση αυτή δύο φορέ ε, κατά τη διάρκεια τη Βελική Προεδρία. Προβλέπονται να γίνουν και άλλε συναντήσει. Είμαι πεπισμένο ότι αν το, το ζήτημα αυτό δεν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια τη ε, Βελική Προεδρία, η επόμενη, η Ουγγρική Προεδρία, θα κάνει ό,τι μπορεί για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Σαστέλ. Οι ερωτήσει 18, 19 και 20 που είχαμε στον κατάλογό μας καταπίπτουν τη απουσία των σύντακτων. Και έτσι σε σχέση με την σύνοδό μας με μια θετική αντιμετώπιση των προϋποθέσεων ότι για πρώτη φορά καταφέραμε σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την ολομέλεια να έχουμε απόλυτη ισότητα μεταξύ των φίλων των Ευρωβουλευτών που είναι παρόντες, παρούσες και παρόντες και έτσι βρισκόμαστε κατά 50% άνδρες και γυναίκες μεταξύ μας. Αυτό είναι κάτι πραγματικά επιθυμητό. Παρότι θα ήταν καλύτερο να διατηρείται αυτή η αναλογία με απόλυτα, απόλυτους αριθμούς και σε μεγαλύτερη αναλογία. Σας ευχαριστώ κύριε Σαστέρ από καρδιάς για τις προσπάθειες και την αποτελεσματικότητά σας. Και θέλω να πω ότι δεν είναι πολύ συχνό όπως συνέβη σε αυτή τη συνεδρίαση σχεδόν όλοι οι συντάκτες να τονίζουν την ε, περιεκτικότητα, την αποτελεσματικότητα των απαντήσεών σας, όπως συνέβη σήμερα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τούτων λεχθέντων τώρα πρέπει να σας αναφέρω ότι θα διακοπεί εδώ η συνεδρίασή μας. Η επόμενη Ολομέλεια θα διεξαχθεί αύριο στις 23 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 12. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λίγη συνεδρίασή μας. Καλό σας βράδυ. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα κυρία Καλή Καληνύχτα αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.